αρμόδια επιτροπή για το θέμα. Η κυρία Μαγδαλένα Άλβαρε τώρα μου ανακοίνωσε γραπτά ότι ορίστηκε αντιπρόεδρο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από 16 Ιουλίου 2010. Το Κοινοβούλιο σημειώνει τον ορισμό αυτό βάσει το άρθρο 7 παράγραφος 1 ε, που έχει να κάνει με την εκλογή ε, ευρωβουλευτών με καθολική ψηφοφορία και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 που ε, κηρύσουν καινή τη θέση αυτή από 16 Ιουλίου 2010. Βάσει του άρθρου 3, παράγραφο